Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία με βάση την απλουστευμένη διαδικασία που αφορά στην έκθεση του κυρίου Ζόντεργκαρτ πρόκειται για την απαλλαγή του 2007. Πρόκειται για τον ε, σχέδιο Δύο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Θα ήθελα λοιπόν να ερωτήσω τον εισηγητή κατά πόσον επιθυμεί να λάβει το λόγο. Διαδικαστικό θέλετε, παρακαλώ. Πρόεδρε, με βάση τον κανονισμό 173 άρθρα 2 θα ήθελα να φερθώ σε δύο κανόνες ε, του ε, κανονισμού μας. Τα μέλη ε, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους με ελεύθερα. Στη συζήτηση σήμερα το πρωί, εσείς κύριε Πρόεδρε,